Uh, um, Κυρίες και κύριοι, μάλλον πρέπει να αρχίσουμε. Έχουμε αρκετούς εμπειρογνώμονες εδώ, στη συνεδρίαση. Καλωσορίζω διακεκριμένα πρώην μας τη Ευρωπαϊκή Κοινοβουλίου, την κυρία Κάρολ Τάγκ, την Κοράτσαν. και έχουμε την έκθεση του... Δεν θα εξετάσουμε το θέμα αυτό γιατί η συνέλεση της του ψηφιακού προγράμματος, ε, της ψηφιακής ατζέντα συνεχίζεται σήμερα και Παύλο Αρίας ε, ξεκίνησε τα εργαστήρια όσον αφορά τη συνέλευση για τα ψηφιακά σήμερα το πρωί στις 9, όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά στο ρόλο του Προέδρου της ομάδας εργασίας μας, όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά και ξέρω ότι σας ε, υποδέχτηκαν καλά. Εγώ εργαζόμουν με τα σκάφη. Λοιπόν, Αυτά που κάναμε στην ομάδα προβληματισμού είναι κάτι που στηρίξαν στις πολιτικές ομάδες. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Και τώρα μπαίνουμε στην... Όλα αυτά εντάσσονται στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Αυτό είναι ανταπόκριση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Έχουμε τον κύριο Λαμότ από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακή Αγορά, που είναι ένας από τους συντάκτες της εκθέσεως και επίσης εκπρόσωπο τη γενική Διευθύνσεως για την Κοινωνία των Πληροφοριών. Λοιπόν, για να ελέγξουμε ποιου έχουμε. Για να δούμε ποιου σκιώδεις έχουμε. Η Εύελιν Γκέρπαρτ είναι εδώ. Εκ μέρου του κυρίου Ντεκάμπο, δεν έχουμε κανέναν άλλον τον κύριο Έμστρομ. Εγώ είμαι σκιώδη για την ομάδα μου. Αν σας αρέσει εντάξει, να σας υπάρχουν αρκετά, αρκετές δουλειές για όλα τα μέλη του ΕΛΚ. Καλωσορίζω όλους εδώ. Α, θα διεξαχθεί μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να παρουσιάσει την ε, έκθεση. Έχουμε ε, μία ώρα για την ε, συζήτηση, οπότε θα καλυφθούν πολλά σημεία. Ο Πάμπλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, συμφωνούμε όλοι από ό,τι φαίνεται. έχουμε και την εκπρόσωπο των σοσιαλιστών που θα εκπροσωπήσει τον κύριο Κορέα Ντεκάμπος. Ε, γνωρίζει ότι, και εγώ γνωρίζω ότι συμφωνεί, γιατί έχουμε ε, συνεργαστεί όλοι μαζί, όχι μόνο με τον ίδιο, ε, αλλά και με τους άλλους σκιώδεις συζητητές. Υπάρχει σχεδόν πλήρης σύμπνοια επί όλων των θεμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σήμερα θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της σημασίας της έκθεσης και των υπολείπων θεμάτων που ε, μας απασχολούν και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο της ψηφιακής αγοράς ε, στην Ένωση. Όλοι τονίζουν τη σημασία του θέματος καθώς επίσης και τις τεράστιες δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη, μεγέθυνση και ε, θέσεις επασχόλησης είναι η ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτό με γεμίζει ικανοποίηση. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά που τώρα αρχίζει και καρποφορεί. Ε, έχουμε εργαστεί σε διάφορες ε, πρωτοβουλίες και προχώρησε πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια προς το κοινό μας στόχο. Μέχρι πρόσφατα δεν γινόταν καν λόγος για την ενιαία ψηφιακή αγορά το θεωρούσαν ε, άπιαστο όνειρο. Γινόταν λόγος για το ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά πάντα σε χρόνο μέλλοντα. Ότι θα ήταν το μέλλον της οικονομίας μας, ενώ άλλα μέρη του κόσμου δρούσαν σε χρόνο ενεστώτα. Γι' αυτό έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ψηφιακή αγορά δεν προχώρησε όσο θα μπορούσε και απέχουμε ακόμα πολύ από την αξιοποίηση όλου του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας. Ε, πιστεύω ακράδαντα και το έχω πει επανειλημμένα εδώ ότι είναι το κλειδί για μια ε, οικονομική ανάπτυξη, τόνωση της κατανάλωσης, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ιδιαίτερα των νέων. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μεγάλος νομικός κατακαιρματισμός που είναι στοιχείο αποτρεπτικό και για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις όταν έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο συνοριακό ψηφιακό εμπόριο. Οι εταιρείε αυτές έχουν να αντιμετωπίσουν 27 σύνορα διαφορετικών κανόνων σε τομεί όπω είναι ο ΦΠΑ, οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε και τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία, για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Γεγονό το οποίο αυξάνει κατά πολύ το κόστο και τα εμπόδια, τα διοικητικά. Τους πιάνει πραγματικός ήλιγκος όταν ε, σκέφτονται ότι πρέπει να αναπτύξουν ε, τη δράση τους σε όλη την Ένωση. Και αυτό είναι απαγορευτικό ιδίως για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν ε, τις δυνατότητες των μεγάλων. Εδώ επανειλημμένα έχουμε πει ότι οι καταναλωτές έχουν μεγάλη αβεβαιότητα και δισταγμό ε, αν θέλουν να αγοράσουν την ψηφιακή αγορά, πόσο μάλλον διασυνοριακή αγορά. Γιατί δεν γνωρίζουν βασικά τις δυνατότητες του μέσου λόγω έλλειψης ενημέρωσης αφενός και λόγω τεράστιας ανασφάλειας δικαίου ακριβώς επειδή είναι κατακαιρματισμένη η αγορά. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα δύο τελευταία χρόνια έχουν αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η δική μας Επιτροπή εργάστηκε πάρα πολύ προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουν εγκριθεί διάφορες εκθέσεις, όπως η έκθεση του 2010, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ή ακόμα και η έκθεση για τα δικαιώματα των καταναλωτών που ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την αύξηση ε, των δυνατοτήτων προστασίας των καταναλωτών online. Έχουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και έχουμε συστήσει και ειδική ομάδα εργασίας για την εσωτερική αγορά. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει και νομοθετικές προτάσεις και αυτό συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό. Και πρέπει να πω ότι εδώ βοήθησε πάρα πολύ η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο τον Ιανουάριο του 2011 που προβλέπει πάρα πολλές προτάσεις και οδικό χάρτη. Δεν θα πρέπει όμως να επαναπαυθούμε στα όσα πετύχαμε, αλλά να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Οι γραμμές που θα πρέπει να δράσουμε είναι διάφορες. Θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τα εξής τρία. Τόνωση της εμπιστοσύνης, ε, αύξηση της ενημέρωσης και προώθηση της καινοτομία. Για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής προσπάθησα να συγκεντρώσω όλες τις απόψεις και τις ε, προτάσεις των σκιωδών εισηγητών στις διάφορες συνεδριάσεις που είχαμε και θέλω να τους ευχαριστήσω για ε, την προθυμία τους και την επικοδομητική τους στάση. Στην έκθεση έχω ε, χωρίσει τη δράση μας σε πέντε μεγάλα μπλοκ ενότητες. Το πρώτο, εισαγωγή αναφέρει τις βασικές γραμμές μια ενιαία ε, ψηφιακή αγορά για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αναφέρω εκεί πέντε σημεία που θα βοηθήσουν στην αύξηση της απασχόλησης σε τέτοιους καιρούς κρίσης που ζούμε. Δεύτερο, τονίζω ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί? Διότι πιστεύω ότι είναι εκ των όνων κάνευ να μπουν στην ψηφιακή οικονομία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό προτείνω τη δημιουργία σχεδίου δράσης για την αύξηση ε, της ενημέρωσής τους νέες τεχνολογίες και να αποκτήσουν οικονομικά και άλλα μέσα για να μπορέσουν να αναπτύξουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα αλλά να έχουν και πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες. Πιστεύω ότι για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί η διασύνδεση των μικρομεσαίων. Αλλιώς δεν μπορούμε να τονώσουμε την κατανάλωση και αν δεν ε, καταναλώνουμε μέσω καινοτομία θα είναι δύσκολο να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση και ανάπτυξη. Αυτή είναι η εξίσωση που φιλοδοξούμε και οφείλουμε να λύσουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 99% των εταιριών είναι μικρομεσαίες και δημιουργούν το 85% των θέσεων απασχόλησης. Οποιαδήποτε ε, πολιτική και πρωτοβουλία για την απασχόληση είναι αναγκασμένοι να περάσουν από τις μικρομεσαίες. Είναι 23 εκατομμύρια οι μικρομεσαίες στην Ευρώπη. Αν αύριο δημιουργήσει έστω και μία θέση εργασίας η κάθε μια, πάει η ανεργία ε, μία νυχτή. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι κλειδί η ψηφιακή οικονομία για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων και για να βοηθήσουμε τις εταιρείες αυτές να βρουν το δρόμο για να βγουν από την κρίση θα πρέπει να τους δίνουμε νέα κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τρίτη ενότητα, αντιμετώπιση των εναπομεινάντων εμποδίων στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Και ζητεί ε, να ξεπεραστεί ο κατακαιρματισμός στο ΦΠΑ τις ε, τραχυδρομικές υπηρεσίες, τις online πληρωμές, στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, οι διακρίσεις βάσει ε, προέλευσης και των καταναλωτών, όλα αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22.2 της Οδηγίας για τις υπηρεσίες. Τέταρτη ενότητα, οικοδόμηση εμπιστοσύνης ε, των καταναλωτών. Η εμπιστοσύνη είναι από τους παράγοντες κλειδιά και μάλιστα τους κομβικούς για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ψηφιακή αγορά θα πρέπει να γνωρίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών με ε, διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου παντού στην Ευρώπη. Περισσότερη ενημέρωση και κατάρτιση διαπαιδαγώγηση, αν θέλετε, των καταναλωτών. Ε, δημιουργία ενός ε, ευρωπαϊκού χάρτη ε, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών. Είναι μερικά από τα μέσα που προτείνω. Και η πέμπτη και τελευταία ανότητα αφορά με τη συγκρότηση της βάσης για μια περισσότερο ανταγωνιστική Ευρώπη. Και τονίζει ότι η ενιαία ψηφιακή ε, αγορά θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα για τις επιχειρήσεις που να διευκολύνει τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη για να έχουν τα εργαλεία εκείνα που θα τους διευκολύνουν το έργο για να μπορούν να υποφελούνται και από ε, την ενιαία ψηφιακή αγορά. Να είναι καλύτερη διασύνδεση και ευρωζωνική πρόσβαση και υπάρχει και ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρχει και η ηλεκτρονική υπογραφή, ε, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπολήθευση. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τις επιχειρήσεις. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ότι πιστεύω ότι η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι για τη μελλοντική της οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να πάρουμε τώρα την απόφαση να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό και όχι εχθρικό επιχειρηματικό κλίμα. Θα πρέπει να δούμε αν είναι η Ευρώπη χωρίς εμπόδια αυτή που θέλουμε, χωρίς φραγμούς. Και φέτος εορτάζουμε την 20η επέτειο της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει να δώσουμε στην οικονομία μας την απαραίτητη όθηση για να δημιουργηθεί μια ουσιαστική ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά στη δεκαετία του 80 και του 90 του περασμένου αιώνα οι τέσσερις ελευθερίες ε, πήραν σάρκα και οστά και αυτό δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες. Σήμερα η διεύρυνση της ενιαίας αγοράς ε, και η επέκταση προς μια ενιαία ψηφιακή αγορά θα αποτελέσει περισσότερες ευκαιρίες και για την οικονομία μας και για τους πολίτες τη δυνατότητα αύξησης απασχόλησης και της ανάπτυξης και της ευημερίας θα πρέπει οπωσδήποτε να δράξουμε την ευκαιρία αυτή και να ξέρουμε ότι μόνο με την απλοποίηση και την έγκριση αυτών των νόμων θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να γίνει πρωταγωνιστής στην παγκόσμια αγορά. Αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό πραγματικότητα, θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς την αντιμετώπιση της κρίσης και η Ευρώπη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Και δεν θα σταματήσω ποτέ να επαναλαμβάνω ότι η έξοδος από την κρίση έχει και ψηφιακή μορφή. Και είναι πολύ σημαντική η στιγμή έτσι ώστε να αρχίσουμε από τώρα τις αλλαγές και την τελευταία διετία που μας απομένει στη θητεία μας να βάλουμε τα θεμέλια για το μέλλον και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αλλιώς θα έχουμε αποτύχει χωρίς καμία αμφιβολία. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σταματώ εδώ και με χαρά να σας ακούσω τους σκιώδης ηγητές και τους υπολείπους βουλευτές της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Παύλο Αρίας. Κάλυψες πολλά σημαντικά θέματα και συμφωνώ μαζί σου. Είναι σημαντική αυτή η ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό την ε, υπογραμμίζουμε και την προσέχουμε. Η κυρία Γκέπχαρτ να δώσει μια πρώτη αντίδραση εκ μέρου του SND. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλιστή. Μα ναι, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ συμβαίνει από καιρού καιρών αυτό. Ο Αντώνιο Κορέγιαντε Αντεκάμπο μου άφησε γαλλικέ σημειώσει, οπότε είναι απλούστερο να μιλήσω γαλλικά σήμερα. Ε, κυριαρίας όπως υποθέσατε και στην αρχή θα πω εν ονόματι του κύριου Κάμπος ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακροσθετική δουλειά ε, πολύ ευχάριστη, σε πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα ο κύριος Κορέα Ντεκάμπος στο σχέδιο εκθέσεως που είναι πολύ ισορροπημένη συμπεριλαμβάνει όλα αυτά που εθίγησα στην ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ομάδα στην οποία συμμετείχε και έκανε μια δουλειά εις βάθος ε, άριστη, θετικότατη. Γενικά, συμφωνεί με αυτά που προτείνατε, αλλά βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία που χρήζουν ε, διευκρινήσεως ή βελτιώσεως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνεί μαζί σας επί των ζητημάτων αυτών. Πρώτα απ' όλα, στο 10 όσον αφορά το θέμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και το πρόβλημα των διασυνοριακών παραδόσεων που συνδέονται με αυτό, όπως και εσείς, δίνει μεγάλη σημασία στο κόστος. Καμιά φορά είναι δυσανάλογο αυτό και ε, εμποδίζει το διασυνοριακό ε, ηλεκτρονικό εμπόριο. Χρειάζεται να είναι αποτελεσματικές οι συνοριακές ε, υπηρεσίες για να εξυπηρετούν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο online. Στο σημείο 11 το θέμα του ΦΠΑ είναι ιδιαίτερο. Το ίδιο ΦΠΑ για τα ψηφιακά και τα φυσικά προϊόντα τα αντίστοιχα είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλα ψηφιακά προϊόντα όπως ο οπτικοκουστικός τομέας και όχι μόνο για τα ηλεκτρονικά βιβλία e-books. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα η ειδική αναφορά στα ηλεκτρονικά βιβλία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής και χρειάζεται διεύρυνση αυτό το πεδίο και είδα από τον τρόπο με τον οποίο γνέφεται ότι συμφωνείτε, νομίζω λοιπόν ότι θα βρούμε σημείο συμφωνίας. Το τρίτο αφορά το σημείο 12, τα μέσα πληρωμών. Θα πρέπει να γίνει εμενία στα νέα μέσα πληρωμών, όπως οι μικροπληρωμές που γίνονται με τα έξυπνα τηλέφωνα smartphones μέσω SMS Εξυπακούεται, εννοείται το κείμενό σας, αλλά ο κύριος Κορέα Ντεκάμπος θα ήθελε να αναφέρεται σαφέστατα και όχι να υπονοείται από το κείμενο. Αυτά τα μέσα πληρωμών θα έπρεπε να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Όσον αφορά το διοικητικό κόστος, που συνεπάγεται κάτι τέτοιο και καμιά φορά μπορεί να είναι αυτό το κόστος μεγαλύτερο από το κόστος της ίδιας συναλλαγής. Άρα θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό και εγώ έχω τέτοια αρκετές, αρκετές παράξενες εμπειρίες σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά τα σημεία 27 με 30, ο Αντώνιο θεωρεί ουσιαστική τη συμπερίληψη στην έκθεση πρωτοβουλίας μιας αναφοράς στην κοινωνική διάσταση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Ε, κυρία Κοράσα Μπίλτ, το ξέρω ότι θα πείτε ότι είναι κανονικό, συνηθισμένο αυτό, εννοείται. Αλλά το, για να έχουμε γενική συνένεση να υπάρχει γενική συνένεση της κοινωνίας, γενική συνένεση να υπάρχει μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων, μεταξύ επιχειρηματιών και εργαζομένων, είναι πολύ σημαντικό θεμέλιο για την ασφάλεια στα κράτη-μέλη και νομίζω ότι πάντα αξίζει τον κόπο να το επενθυμίζουμε. Αναφέρομαι σε αυτό που είπατε σήμερα το πρωί και επιμένω, πρέπει να το πούμε. Δεν αρκεί να λέμε, αλλά συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως στο, στις εργασίες. Πρέπει να το λέμε τακτικά γιατί είναι σημαντικότατο. Αυτό είναι κάτι που προσέθεσα εγώ σε αυτά που έγραψε ο Αντώνιο και σε σκέψη με τις πρωινές σας σκέψεις που εκφράσατε. Και τώρα πάνω σε αυτά που έλεγε Αντώνιο Κορέα, πρόκειται περί αγοράς που θα πρέπει να εξυπηρετεί τους πολίτες και τους καταναλωτές και όλους. Δημόσια υπηρεσία αν θέλετε πρέπει να είναι. Και αυτό είναι σημαντικότατο πέμπτο σημείο που θα ήθελε να θέσει ο Αντώνιο Κορέα Γκάμπους είναι ότι θεωρεί σημαντικότατο να πούμε αν αυτό, αυτό το σήμα εμπιστοσύνης ευρωπαϊκής ε, εξαιρεί τα παιχνίδια online. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πολιτική μας ομάδα και το λέω και προσωπικά. Είναι κάτι που είπα και χτες άλλωστε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν εκεί με τον κύριο Σβάμπ και είπα ότι αυτό το σήμα εμπιστοσύνη για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει μπορεί να δημιουργήσει μια εμπιστοσύνη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι το σημείο σας 24, α, κάτι άλλο το 24. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό και τέλος προτείνει να εφαρμοστεί μια δοκιμή ε, όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπορίο σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία ούτως ώστε να προβλέπονται ποια είναι τα εμπόδια της ψηφιακής αγοράς, να γίνονται δοκιμές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο ίδιος ε, θα αναπτύξει τις σκέψεις του, θα εξηγήσει τι εννοεί όσον αφορά αυτές τις δοκιμές του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτά τα τεστ. Κατηδίαν, πρέπει να πω προσωπικά, διαβάζοντα το κείμενό σας, ότι υπάρχει κάτι που είναι πολύ θετικό, το σημείο 24 όπου υπενθυμίζεται την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διαδίκτυο και τα παιδιά. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικότατο. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που το θίγεται αυτό. Πάνω απ' όλα διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αρμόδια του Κοινοβουλίου, ε, αποφάσισε να μην κάνει έκθεση πρωτοβουλίας επί του θέματος αυτού. Αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Θελήσαμε να συντάξουμε γνωμοδότηση για την ομάδα μας. Περί αυτού πρόκειται, έτσι δεν είναι, Μάλκομ. Ε, είχαμε αποφασίσει να ετοιμάσουμε μια γνωμοδότηση, γιατί κατά την άποψή μα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α εκμεταλλευτούμε λοιπόν το δικό σας κείμενο για να προβάλλουμε κάποια σημαντικά στοιχεία του τομέα αυτού. Είναι ένας τομέας, πιστεύω, πολύ ουσιαστικός και δεν νομίζω ότι μπορούμε να λέμε απλώς ότι ανησυχούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια ανακοίνωση, εντάξει, τελεία και παύλα. Νομίζω ότι αυτό είναι αξιοθρύνητο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βασιστούμε στην έκθεση πρωτοβουλία σας σαν βάση για να στείλουμε κάποια σημαντικά πολιτικά μηνύματα σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Ε, Όλος ο κόσμος μιλάει γαλλικά σήμερα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αλλά καλύτερα εγώ να τα πω αγγλικά. Θα είναι δύσκολο γαλλικά. Εγώ θα μιλήσω εκ μέρους της ομάδος μου και μετά φαντάζομαι ότι και η κυρία Γκάλο και η κυρία Κοράτσαμπίλ θα ήθελαν να πάρουν το λόγο και ο κύριος Φαμπ. Όλοι μπορείτε να πάρετε το λόγο. Καταρχά. συμφωνώ ότι ο Παύλο Αρία ε, εκπώνησε μια πάρα πολύ καλή έκθεση που επικεντρώθηκε σε πολλά σημαντικά ζητήματα γιατί ένα τμήμα της σημαντικής δουλειάς που προσπαθούμε να κάνουμε και έχουμε κάνει και με την ε, ε, πράξη της ενιαίας αγοράς Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο πολύ συνεκτικοί, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σφαιρικοί στην προσέγγιση μας ε, άλλωστε αυτό είπε και ο Μισελ Μπαρνιέ σήμερα το πρωί. Χρειαζόμαστε, έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας ε, και είναι και θέμα προστασίας δεδομένων που είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε επίσης και θα έχουμε και εκεί τη δυνατότητα να ε, συζητήσουμε το ε, σημείο αυτό. Μπορούμε ούτως ή άλλως ε, στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων θα συζητήσουμε ορισμένα πράγματα που αφορούν την ενιαία ψηφιακή αγορά και μάλιστα μερικά δύσκολα, περίπλοκα ζητήματα γιατί σε μερικές ε, χώρες ε, υπάρχει, υπάρχουν συναλλαγές online, αγορές online, γιατί ακριβώς ε, υπάρχουν επαρκείς και αξιόπιστες παροχές της δυνατότητας αυτής και μάλιστα καμιά φορά σε τιμές πολύ καλές Νομίζω ότι ειδικότερα οι αγορές στο διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι μια σημαντική εμπειρία για τους πολίτες. Ε, δίνει τη δυνατότητα ε, η αγορά στο ίντερνετ ε, στους εμπόρους να παρέχουν πολύ δικευμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένα προϊόντα σε τεράστιες αγορές. Ειδικευμένα προϊόντα λοιπόν παρέχονται με αυτόν τον τρόπο και έτσι οι ε, έμποροι μπορούν ε, να δραστηριοποιούνται σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη, στο φόρουμ Ενιές αγοράς στην Κρακοβία Θυμάμαι ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που ετέθησα ήταν μια μικρομεσαία επιχείρηση που ε, ήθελε από την Αυστρία να, ε, να, ε, να πουλήσει ένα είδος φρουτοχυμού ή τέλος πάντων κρασιού από φρούτα στην Γερμανία και είπε ότι υπήρχε επιπλέον κόστος μεταφοράς στην Γερμανία από την Αυστρία. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια τέτοια ζητήματα απλά, ε, τα ζητήματα διανομής, τα οποία ε, είναι πολύ σημαντικά και μπορούμε να επικεντρωθούμε στο να είναι πιο ε, ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας, αλλά παράλληλα να, υπάρχουν, να υπάρχει και ενημέρωση για τους καταναλωτές μας. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρξουν παράλληλα. Η ενιαία ψηφιακή αγορά αφορά και αυτό το θέμα ε, τα ψηφιακά μέσα μας δίνουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Λέμε συχνά ότι επειδή είναι ψηφιακό κάτι είναι καινούριο και διαφορετικό. Όμως ε, κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές και τους αγοραστές ε, είναι ζητήματα που υπήρχαν ούτως ή άλλως και εκτός διαδικτύου. Άλλωστε ε, πρέπει να θυμόμαστε και τον τίτλο ε, «Το συνεκτικό πλαίσιο» έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για το θέμα αυτό. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο κάπως το έχουμε ξεχάσει σε σχέση με τη δημιουργία της ενίας αγοράς, γιατί μας ενδιαφέρει η τεχνολογία, αλλά πρέπει να δούμε και τα βασικά εργαλεία με τα οποία ε, εξυπηρετούμε τους καταναλωτές μας. και έχει να κάνει και με, απολύτως με τη στάση των καταναλωτών ε, όσον αφορά τις, ε, ε, τις, αγοράς, τις αγορές στο ίντερνετ. Εγώ τα λέω όλα αυτά για να τονίσω ορισμένα ε, στοιχεία που ούτως ή άλλως ανέφερε και ο Πάμπλο. Κάτι ακόμη, η πληροφόρηση των καταναλωτών στο πλαίσιο της εμπιστοσύνης είναι και αυτή ε, σημαντική. Έχει σημασία από πού αγοράζουν, πού βρίσκεται η εταιρεία και πού θα απευθυνθούν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα οι ε, καταναλωτές. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ισχύει πάντοτε, ε, δεν εφαρμόζεται σωστά η ισχύουσα νομοθεσία και οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί που μπορεί να έχει κάποιος πελάτης με κάποιον προμηθευτή είναι πάρα πολύ Είναι, είναι, είναι ε, σημαντικό τμήμα των μηχανισμών αυτών. Γι' αυτό Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά και η πρόταση όσον αφορά το πρόγραμμα των καταναλωτών ε, εξετάζει ακριβώ αυτό το θέμα. Μπορεί να μην έχετε δει τις λεπτομέρειες. Ε, το σύστημα πληροφοριών της ε, εσωτερική αγοράς που το εγκρίναμε σήμερα το πρωί αφορά ακριβώς και την ε, οδηγία του ηλεκτρονικού εμπορίου που πρέπει να είναι τμήμα όλου αυτού του πλαισίου και είναι σημαντικό για να συμπληρωθεί η εικόνα και πρέπει να ε, επικεντρωθεί και η προσοχή των κρατών μελών στην εφαρμογή των σχετικών ε, κανόνων. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα το, βλέπ, το οποίο βλέπουμε στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τα ζητήματα των προγραμμα, του προγράμματος των καταναλωτών. Υπάρχουν κάποιες ιδέες για την κατάρνηση, για τις δεξιότητες των προμηθευτών στο διαδίκτυο σε σχέση με τις δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Ε, να υπάρχουν προγράμματα ανάπτυξης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη αλλά πρέπει επίσης και ολόκληρη η πτυχή των καταναλωτών να συμπεριληφθεί. Ε, όταν συζητούσαμε, όταν, όταν κάναμε ένα, μια, ένα πολύ σημαντικό ε, εργαστήριο για την ψηφιακή οικονομία, συμμετείχαμε με, ε, συμμετείχαν οργανώσεις καταναλωτών με, με, με τις οποίες συζητήσαμε και είδαμε με ποιους τρόπους μπορούμε πολύ απλούστερα να παρουσιάσουμε τα δικαιώματά τους στους καταναλωτές, γιατί υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα υπό την οδηγία των, ε, για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, και πέραν ε, από την συζήτηση που αφορά το, ε, τον, την ομοθεσία για τις πωλήσει, ίσως θα πρέπει να έχουμε και έναν κώδικα δεοντολογίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η αφετηρία αυτή, γιατί έξι από αυτά τα σημεία ούτως ή άλλως υπάρχουν στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν ε, λέμε τίποτε καινούριο, ε, ούτε αναφέρουμε κάτι καινούριο, απλώς ε, επικεντρώνουμε την προσοχή στην εφαρμογή των, της οδηγίας αυτής. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μεταγράψουν τα στοιχεία αυτά και μάλιστα πολύ σύντομα, ώστε να είναι στη διάθεση όλων. Άλλα στοιχεία του κώδικα ε, πρακτικής ε, θα αφορούν ε, τον τομέα των λιανικών πωλήσεων και τις καλές πρακτικές στον τομέα αυτό, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι όλα Το trust marks, τα trust marks είναι πάρα πολύ σημαντικά μεν, αλλά δεν υπάρχουν ε, πάντοτε ως τμήμα των ε, διαδικασιών και των, του πλαισίου που προσπαθούμε να θέσουμε. Χρειάζονται όμως προώθηση, ενθάρρυνση, ε, γιατί διαφορετικά αν δεν αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές, αν ένας έμπορος έχει ένα συγκεκριμένο τέτοιο σήμα, πρέπει να έχει αξία και για τον ίδιο τον έμπορο. Υπάρχουν ε, οικονομίες ε, ε, κλίμακας, οι οποίε θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν προ αυτήν την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι ένα τμήμα της δουλειά για τη στρατηγική της λιανικής αγοράς, τη οποία ηγείται η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, έχει άμεση σχέση με αυτό και είμαι σίγουρο, ότι θα πει κάτι γι' αυτό στη συνέχεια. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να μην το ξεχνούμε. Το θέμα των πληρωμών επίσης, που ακόμη το επεξεργαζόμαστε, το έχουμε ήδη αναφέρει, Υπάρχει μια σαφής αναφορά εδώ που έχει να κάνει με τα ζητήματα ε, των φαρμακευτικών προϊόντων, των φαρμάκων που ε, υπάρχουν στο διαδίκτυο και πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό. Πολλές ε, απόψεις ακούμε από τις διάφορες επιτροπές και η Επιτροπή Λίμπε και η Επιτροπή Πολιτισμού Νομίζω όμω ότι κυρίω με του συναδέλφου τη Επιτροπή Περιβάλλοντο πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν ε, προβλήματα όλο και περισσότερα που έχουν να κάνουν με παραποιημένα φαρμακευτικά προϊόντα ε, και αυτό μας φέρνει και στο ευρύτερο πρόβλημα της παραποίηση. Κάτι ακόμη. Ναι. Κάτι ακόμη είναι ότι υπάρχουν και κάποια εργαλεία στο πλαίσιο των πακέτων τηλεπικοινωνίας, ε, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Όταν ε, μιλήσαμε για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ε, ένα θέμα για το οποίο εγώ ήμουν εισηγητής, ένα από τα πράγματα που ε, εισαγάγαμε για πρώτη φορά ήταν η δυνατότητα υποχρέωση των παρόχων ίντερνετ στα κράτη-μέλη να στέλνουν ένα μήνυμα σε όλους τους καταναλωτές τους και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ήταν ο κίνδυνος για τα παραποιημένα φαρμακευτικά ε, προϊόντα ή ας πούμε για τη χρήση του ίντερνετ από τα παιδιά, για την ασφάλεια στο ίντερνετ, όπως επίσης και για την ασφάλεια του υπολογιστή. Δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος ε, ε, δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο η υπεύθυνοι ρύθμιση των ε, ε, τηλεπικοινωνιών είναι σε θέση να εντοπίσουν ε, οποιαδήποτε παραποίηση οποιαδήποτε λάθος χρήση του ίντερνετ, αλλά ούτως ή άλλως όλο και περισσότερα τα ζητήματα των, της προστασίας των καταναλωτών σχετίζονται με αυτό το πακέτο των, των τηλεπικοινωνιών. Εντός ή άλλως γίνονται και συγκρίσεις τιμών που θα έπρεπε να επεκταθούν και σε άλλα ζητήματα βέβαια. Κάτι ακόμη, θα συζητήσουμε για την ε, προστασία δεδομένων, θα τα ξαναπώ ενδεχομένως τα ίδια πράγματα, αλλά θα τα πω και τώρα. Υπήρχαν ε, κάποιες διατάξεις ε, στο, στην προστασία του, στο e-privacy, το οποίο αφορούσε ακριβώς το κατά πόσο θα αποκαλύπτονται κάποια δεδομένα που αφορούν τις ε, συναλλαγέ και νομίζω ότι πάλι έχει να κάνει με την οδηγία προστασίας δεδομένων ε, και επίσης παρατήρησα ότι τα νέα σχόλια που αφορούν ε, το γεγονός ότι οι ιστότοποι δίνουν πληροφορίες για τους κανόνες λειτουργίας τους και τις προδιαγραφές τους, ε, για ε, τα cookies για παράδειγμα που αφορούν τις συναλλαγές, εμφανίζονται όλο και περισσότερο στον ιστότοπο και αυτό είναι αποτέλεσμα του τι εγκρίναμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Και ε, το λέω αυτό σε σχέση με την διαδικασία ε, των σχετικών οδηγιών, τις οποίες επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Για μένα είναι σημαντικό αυτό το ε, κείμενο γιατί ε, συγκεντρώνει πολλά στοιχεία που αφορούν διάφορους τομείς και δίνει, δίνει μια πολύ σφαιρική εικόνα και τονίζει, συνδέει διάφορες, διάφορες διαφορετικές πτυχές μεταξύ τους. Και νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση αυτή για να κάνουμε... να, να κάνουμε μια πολύ σφαιρική δήλωση και για την ε, εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών, των πελατών μας. Αυτή η εμπιστοσύνη σημαίνει βέβαια και καλύτερες συναλλαγές για όλους. Αυτή είναι η δική μου ε, συνεισφορά εκ μέρους του ε, σκιώδου συζητητούς μου. Η Άννα Μαρία φαντάζομαι θέλει να πάρει το λόγο. Sorry. Κοιτάξτε, θα βάλω όλους τον κατάλογο αγορητών και όποιο θέλει να αρνηθεί, να συμπεριληφθεί, μπορεί να το κάνει. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, λοιπόν. Ευχαριστώ, όλα τα είπατε. Τα είπε όλα, Μάλκομ. Πάμπλο. είναι πολύ καλή αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται να περάσει αυτή η ατζέντα ψηφιακή. Στην έκθεσή σου και στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε μια βάση για να προχωρήσουμε. Θέλω να πω ότι θα έπρεπε να κινηθούμε επιγόντω για να εφαρμόσουμε το ψηφιακό αυτό πρόγραμμα, την ψηφιακή ατζέντα. Πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει οδικό χάρτη, δηλαδή χρονοδιάγραμμα για τις διάφορες δράσει, αυτέ που αναφέρονται είναι ένα ευρύ φάσμα πρέπει να καλυφθεί και χρειάζεται μια συνοχή. Να πούμε τι θα κάνουμε και πότε. Στην παράγραφο 3. Είναι το βήμα. Το άλλο. Από την εμπειρία που έχω, έχοντας δημιουργήσει μια εταιρεία το 99 ηλεκτρονικού εμπορίου και επί σειρά ετών πριν πω στο κοινοβούλιο την διοικούσα, ε, υπήρχαν πολλά πρακτικά προβλήματα. Ένα επιχειρηματίας σαν και εμένα αισθανόταν τον εξαπατούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω αυτό. Μου λέγανε μπορεί να πωλήσει αγαθά διασυνοριακά στο διαδίκτυο. Επιτρέπεται. Και είχε γίνει μεγάλη εκστρατεία που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έλεγε, ξεκινήστε, κάντε το. Στην πράξη χτυπά το κεφάλι σου, λόγω κατακαιρματισμού. Δεν, θέλω να επαναλάβω αυτά που έλεγε. Ε, πολλά από αυτά που είπαν και συνάδελφοι την άλλη πλευρά μα βρίσκουν συμφώνου. Το θέμα του κόστους διανομής, το έζησα, μεταφορών και παράδοσης είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα. Το 2012 έχουμε τέσσερις πολυεθνικές που κυριαρχούν στην αγορά για τις διασυνοριακές πωλήσει. Τεράστιο κενό μεταξύ κάποιων κρατών μελών. Σε κάποια κάτι μέλη είναι πολύ ανταγωνιστικό στο μέσα, αλλά καθόλου. Δεν είναι μόνο το κόστος. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς μια εταιρεία η οποία θα διανέμει τα αγαθά σου από Ιταλία στη Σουηδία, Φερρυπίν που να παρέχει μια υπηρεσία, να παραδίδει τα προϊόντα Σάββατο, Κυριακή, μετά τις 6 το απόγευμα. Σε μια χώρα όπου εργάζονται οι περισσότεροι όλοι μέλα, περιορίζεις την αγορά αν μπορείς να παραδώσεις μόνο Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και μέχρι 6 το απόγευμα. Λεπτομέρεια φαίνεται, αλλά ήδη αφήνει πολλούς εκτός αγοράς. Σχεδόν όλους όσους εργάζονται. Και πρέπει να πας σε εθνική εταιρεία για τη διανομή και αυτό αυξάνει το κόστος. Μετά είναι το θέμα του, της εφορίας, των φόρων. Δεν είμαι υπέρ φορολογικής εναρμόνισης, αλλά ένα τιμολόγιο για κάτι... Περνάει για κάτι που πολλέ μπορεί να έχει 4 ΦΠΑ αν περνάει από χώρε. Και πρέπει να έχεις καταχωρήσει την εταιρεία για το ΦΠΑ και να το δηλώσει στη χώρα ε, Έδρα της εταιρεία και στην χώρα του πελάτη. Πρέπει να έχεις λογιστές και στην έδρα σου, στη χώρα έδρας και στην μεγαλύτερη αγορά πελατών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με εταιρείε που μπορούν να έχουν διπλά λογιστικά. Δύο λογιστές αν θέλετε. Ε, και αυτό είναι πολύ μεγάλο διοικητικό κόστο. Γι' αυτό καλωσορίζω την ιδέα των δοκιμών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το είχα προτείνει. Ό,τι αποφασίσουμε σε άλλου τομεί να έχουμε υπόψη μα πώ επηρεάζεται η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Από τη δική μου εμπειρία τι είδα. Ω διαμόρφωση πολιτική επικρατούσε μια ιδέα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι απειλή για το εμπόριο. Άρα χρειάζονται ξεχωριστοί κανόνε για να το κρατούν εκτό. Αλλά αυτό που έθεσε επιτάπητο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι άλλο ότι ίσως πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπληρώνει το εμπόριο. Είναι μια δυνατότητα, δυναμικό, δυνατότητα να αυξηθούν, να αναπτυχθούν οι μικρές εταιρείε, να χρησιμοποιούν περισσότερα μέσα και να ανταγωνίζονται δυσυνοριακά χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και του καταναλωτέ από μακρές περιοχέ κλπ. να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε που δεν θα είχαν διαφορετικά. Αυτό είναι αλλαγή νοοτροπία του πώ βλέπουμε το εμπόριο και θα πρέπει και συγκεκριμένα μέτρα να μεταφραστεί αυτό, γιατί για την ώρα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Λίγα πράγματα. Το γενικό θέμα του διαδικτύου. Πρέπει να το εξετάσουμε και να το αντιμετωπίσουμε τις πωλήσει μέσω διαδικτύου με τον ίδιο τρόπο και αξιοπρέπεια όπως το κανονικό εμπόριο. Και η ουδετερότητα σαν αφορά την νομοθεσία είναι κάτι σημαντικό. Μετά, το άλλο που έθεσε ο Μάλκορν που με ενδιαφέρει πολύ. Το ασφαλές διαδίκτυο για τα παιδιά. Στην παράγραφο 24 αναφέρεται το θέμα των διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Η ελευθερία του διαδικτύου είναι υπέροχη και για τα παιδιά. Τους δίνει δυνατότητα για παιδεία, για επικοινωνία κλπ. Όμως θα πρέπει να έχεις επαφή με τους επιχειρηματίες για τι υπεύθυνε διαφημίσει, τι προσεκτικέ διαφημίσει στο διαδίκτυο. Υπεύθυνοι πολιτικέ διαφημίσει. Και ξέχασα και κάτι για το διαδίκτυο. Το ανέφερε και ο Μάλκομ για το τεχνικό εμπόριο. Το θέμα τη ενημέρωση. Εφόσον δεν υπάρχουν η ετικετοθεσία και σήμανση, όπω σε ένα κατάστημα, δεν μπορεί να διαβάσει στο διαδίκτυο την ετικέτα του προϊόντο, και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να δώσουμε δυνατότητα στους καταναλωτές να μην συγκρίνουν μόνο τιμές αλλά και ποιότητα. διαθέτοντας και προβάλλοντας τις ε, κατάλληλες πληροφορίες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο κ. Χάρμπορ. Αυτό για το φόρο μου θυμίζει ότι είμαστε σημείο μας και ο συγκητής και αυτό που έπρεπε να αναφέρω ήταν ότι υποστηρίζουμε μεν οι διαδικασίες του VAT κάπως να εναρμονιστούν, δεν είμαστε όμως Θέλουμε οι διαδικασίε του ενίσπραξη του ΦΠΑ να ευθυγραμμιστούν και να συντονιστούν, αλλά δεν θέλουμε εναρμόνιση του ΦΠΑ. Η ε, κυρία Γκαλό, έχει το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώ. Τρει παρατηρήσει έχω να κάνω. Θα αρχίσω από μια παρατήρηση για τη φορολογία. Τονίζοντα ότι δεν πρόκειται τόσο για εναρμόνιση, αλλά για να μπορούν τα πολιτιστικά αγαθά, ας πούμε, online να υπόκεινται σε χαμηλότερο ε, συντελεστή ΦΠΑ όταν ισχύει το ίδιο ε, για ε, το προϊόν αυτό καθ' αυτό. Μπορεί να είναι βιβλία, δίσκοι κτλ. Δεν τίθεται εδώ θέμα κινδύνου εναρμόνιση. Θυμίζω ότι σε σχέση με αυτό το κοινοβούλιο, ναι, είναι γεγονός, κατόπιν δικής μου πρωτοβουλίας ψήφισε ψήφισμα με πλειοψηφία 484 ε, ψήφων υπέρ και τώρα είναι ε, κάτι που εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις, αλλά το Κοινοβούλιο την κατάλαβε αυτή την ανάγκη. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω. Δεν θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο οι καταναλωτές στην ανάπτυξη αυτής της ψηφιακής αγοράς, αλλά και όσοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, όπως είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γιατί είναι προφανές ότι για να πληρώνεις, για να γράψει συνδρομητή, υπάρχουν κάποιε διαδικασίε οι οποίε θα πρέπει και αυτέ να εξελίσσονται όσο εξελίσσεται και το εμπόριο. Και Επίση, τολμώ να πω ότι οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε δεν είναι πάντα στο ύψο των περιστάσεων. Αυτοί οι δύο εταίροι πρέπει επίσης να συμμετέχουν τουλάχιστον εξίσου με ε, τις οργανώσεις των καταναλωτών. Και μια τρίτη παρατήρηση αφορά ένα θέμα που θα έχουμε το χρόνο, άπλετο χρόνο να συζητήσουμε και είμαι εγώ η συγγήτρια, η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει και εκεί να είμαστε άκρος προσεκτικοί και να μην αφαιθούμε, όπως κάνουμε κάθε φορά όταν πρόκειται για το διαδίκτυο, να μας παρασύρουν σε μια τελείως τρελή ιδεολογία. Να προστατεύονται τα πάντα απολύτως ε, σε βαθμό που να είναι τροχοπέδι για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εκεί θα πρέπει να βρούμε τη λεπτή ισορροπία. Να είμαστε λιγότερο ιδεολόγοι, περισσότερο πρακτική και αν θέλουμε να αναπτύξουμε πραγματικά αυτό το ηλεκτρονικό εμπόριο θα χρειαστεί να εκτιμήσουμε στη σωστή διάσταση αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες που είναι τόσο ανεπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι και τόσο μη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή να το έχουμε και αυτό υπόψη μας αν θέλουμε να πετύχουμε. Και επίσης το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει εμείς να προνοούμε, να προτρέχουμε. Και όχι μόνο αυτό, είναι και το θέμα του cloud computing. Και είναι και αυτά θέματα τεχνολογίας και τεχνολογικής εξέλιξης. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιο άλλο. Και Σφάμπ. Η κυρία Βερχάιεν πρώτα. Οι κυρίε πρώτα προηγούνται. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του που είναι εκτενέστατη. Με την ψηφιακή ατζέντα πραγματικά έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα και αφορά το διαδίκτυο και διάφορες υπηρεσίες. Αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε κάτι που θα μας απασχολήσει και στα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης ότι θα πρέπει να έχουμε και την απαραίτητη υποδομή κάθε φορά και για τις μικρομεσαίες ακριβώς επιχειρήσεις ε, στην Ήπεθρο να μπορούν να εποφελούνται από μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή αγορά. Θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να τα συμπεριλαμβάνουμε στη στρατηγική μας γιατί να μην έχουμε στην Ευρώπη μια κοινωνία δύο κατηγοριών ή ταχυτήτων, από τη μια τα μεγάλα αστικά κέντρα που έχουν ήδη τις υποδομές και από την άλλη ύπεθρος που ε, θα εποφεληθεί καλύτερα ακριβώς και ο ιδιώτης καταναλωτής της υπέθρου από αυτή τη δυνατότητα ηλεκτρονικού εμπορίου. Ε, αλλά θα πρέπει να έχουν και την πρόσβαση. Θα πρέπει να λύσουμε κάποια προβλήματα Πολλοί συνάδελφοι τα ανέφεραν, είναι και τα φορολογικά, είναι η προστασία των δεδομένων, πώς μπορώ να εξασφαλίσω προστασία και ασφάλεια των ε, καταναλωτών χωρίς να αποκαλύψω πάρα πολλά πράγματα, αλλά να γνωρίζω ένα την ταυτότητα του άλλου. Ποιος είναι αυτός που μου πουλάει, ποιο είναι αυτός που αγοράζει. Γιατί το διαδίκτυο σήμερα ε, αναπτύχθηκε σε μια πολύ φιλελεύθερη δομή, ή θα υπάρχουν όμως και κανόνες. Να δημιουργηθεί εκεί το ηλεκτρονικό εμπόριο που ακόμα δεν υπάρχει και να υποφελούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Mr. Schwab. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να το πω ως εξής. Δεν θα απαντήσω σε όλα όσα ήθελα να πω, ε, ακόμα και αν είμαι τελευταίος, γιατί δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα, ούτε χρειάζεται να τα επαναλάβω. Είναι πολύ καλή η έκθεση. Ε, όλα τα υπόλοιπα τα είπαν οι προλαλήσαντες ή τα έχει καλύψει ο ίδιος ο εισηγητής τόσο λαμπρά που δεν χρειάζεται εγώ να τα αναφέρω. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στο σημείο 10 που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ζητάει να βρει λύσεις για τη βελτίωση λέει, του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις υπηρεσίες παράδοσης ε, προϊόντων που αγοράζονται ηλεκτρονικά. Συμφωνώ, αλλά τι σημαίνει αυτό. Ότι μέχρι τώρα είχαμε κάποιες εθνικές ρυθμίσεις, το είπε τώρα η Σαμπίνε Φερχάη, για να εξισορροπούν την κατάσταση μεταξύ αστικών και ε, υπαίθριων αγροτικών περιοχών. Τι θα γίνει δηλαδή η ε, υποδομή ε, και οι υπηρεσίες των ταχυδρομείων θα γίνουν από εθνικές, ευρωπαϊκές και θα υπολογίζεται και το κόστος αντίστοιχα. Δεν είναι εύκολο γιατί μέχρι τώρα το ταχυδρομείο είχε εθνικό μονοπόλιο ή θεωρείται κοινοφελής υπηρεσία γιατί θα πρέπει να φτάνει το ταχυδρομείο σε κάθε σημείο της επικράτειας μια χώρα. Είναι τόσο εύκολο, δεν νομίζω, δεν είναι τόσο απλό ε, αυτό οι εθνικές ε, ταχυδρομικές υπηρεσίες να γίνουν ευρωπαϊκές. Αλλά όταν μιλάει ο εισηγητής για ενιαία τιμή ε, παράδοσης και αποστολής, έχει να κάνει με αυτό. Θέλω επίση να αφαιρθώ σε ένα άλλο σημείο στο 17 και χαίρομαι που ο συνάδελφος Άριας εδώ αναφέρεται στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και ζητάει κάποιον εναρμονισμό και να φροντίσουν τα κράτη-μέλη να ε, εφαρμοστεί αυτό, λέει να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της. Έχει δίκιο. Αλλά αυτό ισχύει και για την έκθεση για τη λεγόμενη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Και θα πρέπει να το κοιτάξουμε προσεκτικά αυτό. Γιατί στη χώρα που γνωρίζω εγώ και έχω εκλεγεί, τι γίνεται. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει εφαρμόσει σε ένα πρώτο βήμα ε, αυτά τα μέσα που ζητάει η οδηγία και τα, και τα πρόβαλε ως δικιά της ιδέα και ποια ήταν αυτά τα θετικά για τους καταναλωτές. Το υπόλοιπο ε, έρχεται και αυτό να το εφαρμόσει και λέει ότι αυτό μας το επιβάλλει η Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να έχουμε συμβιβασμούς όμως για όλη την Ευρώπη και να είναι ε, η μέση οδός. Και τα κράτη-μέλη ε, τελικά θα υποχρεωθούν με ένα σπάρο να πάρουν όλα τα μέτρα έτσι ώστε ο χαρακτήρας του συμβιβασμού που έχει επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ε, είναι σαφής και να ισχύει για τους πολίτες σε κάθε χώρα μέλος. Αυτά ήθελα να πω, τα άλλα τα υποστηρίζω, υπόθηκαν ήδη, δεν θέλω να τα επαναλάβω και ελπίζω η έκθεση Άριας να γνωρίσει ευρία πλειοψηφία τελικά. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει. Καλώς. Θα ζητήσω την πατήσει Αλαμότ αν θέλει να σχολιάσει τα όσα άκουσε μέχρι τώρα και αν θέλει να πει κάτι άλλο. Και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Αρίας για να συνοψίσει και θα καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στην ποιότητα της εργασίας του εισηγητή για το θέμα αυτό, αλλά γενικά και την δουλειά των συναδέλφων στις ομάδες εργασίας που έχουμε παρακολουθήσει εδώ και δύο χρόνια. Βλέπουμε τη σύγκληση απόψεων που μας εκονοποιεί ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Επιτροπής σας, αλλά και ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο, γιατί για το θέμα αυτό, δεδομένου των συμπερασμάτων ε, στα τέλη Μαρτίου του ε, Συμβουλίου και περιμένοντας να δούμε τι θα πει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, ελπίζουμε ότι ε, η ψηφιακή αγορά θα είναι αναγνωρισμένη από όλους. Για ορισμένα ζητήματα τα οποία θέσατε, καταρχάς σημείωσα τις προτεραιότητες που αναφέρατε Ειδικότερα ε, σημείωσα το θέμα ε, των, ε, της διανομής και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Γνωρίζετε ότι είναι μία από τις μεγάλες προτεραιότητες που έχουμε για τα επόμενα έτη, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα πρόσκομα στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μας είπατε πόσο δύσκολο είναι το θέμα. Ε, θα είναι και δύσκολο να βρούμε λύσεις. Θα αρχίσουμε μια μεγάλη διαβούλευση στο τέλος αυτής της χρονιάς όμως είναι γεγονός ότι είναι ένα ε, δύσκολο θέμα, απαραίτητο όμως. Για το ΦΠΑ επίσης ε, άκουσα τα αιτήματά σας ε, για ουδετερότητα του φόρου μεταξύ των ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών αγαθών. Υπάρχει ένα ζήτημα για το μέλλον των καθεστώτος του ΦΠΑ. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα του οποίου επικεφαλής είναι ο Επιτροπός ΕΜΕΤΑ και νομίζω ότι θα έχουμε σύντομα απαντήσεις. Και για το θέμα τώρα του, της δοκιμής ε, του ψηφιακού εμπορίου, του e-commerce που αναφερθήκατε και εσείς, ήταν μια ιδέα την οποία ε, είχε προταθεί στο πλαίσιο των συμπερασμάτων της ανακοίνωσης ε, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματά σας, θα δούμε τώρα εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορούμε να ε, επισημοποιήσουμε αυτήν την δοκιμή ώστε να ε, βεβαιωθούμε ότι ε, ανταποκρίνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος Παύλο Αρίας, τα συμπεράσματά σας. Gracias a todos los que eh, han participado en este debate. Eh, yo he tomado también muy buena nota de todos los temas. Eh... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σημείωσα και εγώ όλα τα θέματα και σε γενικές γραμμές συμφωνώ πάρα πολύ με όλα αυτά που ακούστηκαν. Αλλά επίσης ισχύει ότι το κείμενο, ξέρετε, έχει περιορισμό χαρακτήρων. Ε, δεν μπορεί να είναι πολύ μακροσκελές, γι' αυτό ε, περιορισμένοι στην έκφρασή μας και είναι και σχέδιο ίδιας πρωτοβουλίας, καταλαβαίνετε και ξέρετε ότι είναι περιορισμένο το εύρος ε, της έκθεσης. Με τις τροπολογίες ίσως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο με τον τρόπο που ακούσαμε και είμαι στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε. Τα σημείωσα όλα αυτά. Το, το θέμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών πραγματικά κυριαρχεί σε αυτή την ανταλλαγή και ε, νομίζω ότι πράγματι αυτά τα θέματα θα μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε με τροπολογίες. Αυτά. Πρόεδρε, να πούμε λίγο τα χρονοδιαγράμματα τώρα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 10 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, 10 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι και από εκεί και πέρα θα δούμε τις τροπολογίες και θα προχωρήσουμε γιατί είναι τα βασικά θέματα αυτής της ιτίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Yes, that's right. The 10th of July. Μάλιστα. 10 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε γέρος ε, στις 18 Σεπτεμβρίου τις ε, μεταφράσεις. Θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Σίγουρα θα γίνει κάτι τέτοιο και μετά θα ψηφίσουμε 11 Οκτωβρίου και ελπίζω ότι θα σεβαστούν το χρονοδιάγραμμα αυτά όλες οι γνωμοδοτούσες επιτροπές. Ε, ελπίζω να θεωρήσουν ε, το σύντημα διανομή και, οι, και άλλες επιτροπές, κυρίως η Επιτροπή Μεταφορών ως σημαντικό ζήτημα. Ε, το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα στο εργαστήριό μας και ε, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μας απασχολεί πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Λαμό, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον εισηγητή. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γιατί όλα τα ψηφιακά μιλάμε σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση της κυρίας Γκάλο για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών. Θα κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία των δεδομένων ε, πρώτα. Ενημερωτικά να σας πω ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, που είναι η αρμόδια επιτροπή, συζητά την ενισχυμένη συνεργασία δεν έχει ακόμα επιληθεί το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, εμεί θα συνεχίσουμε με τη δική μα έκθεση. Γιατί ξέρω ότι η Επιτροπή ε, Ελευθεριών του Πολίτη έχει πάρα πολλέ διαβουλεύσει αυτή τη στιγμή με ε, του φορεί ελέγχου προστασία των δεδομένων στα διάφορα κράτη-μέλη και καλό είναι να μην καθυστερήσουμε κι εμεί. Είναι καλό λοιπόν να συνεχίσουμε τη δουλειά μας ε, και θα δούμε η Λάρα ακόμη τι έχει να μας πει. Η κυρία Σαλντεμόζο δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα το απόγευμα. Κρίμα. Λάρα, μόνη σου είσαι λοιπόν. Ελπίζω να έχουμε σχόλια και από τους υπόλοιπους. Εγώ θα σου πω την, την άποψή μου ούτως ή άλλως. Φαντάζομαι το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ας αρχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση για την προστασία των δεδομένων. Λάρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια συντομότατη αναφορά σε αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελευθεριών διότι είμαστε στενή επαφή, στενή συνεργασία ακριβώς για να μην μένουμε πίσω όσον αφορά τη δραστηριότητα και είναι ένα από τους λόγους για τον οποίο ζήτησα να παρατείνουμε ε, την προθεσμία για τις 12 για το σχέδιο κειμένου διότι θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές ή πρωταγωνιστές στον τομέα αυτό θα ήθελα να πω ότι για μία ακόμη φορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επιβεβαίωσαν το ότι θέλουν να πλησιάσουν τους πολίτες, κυρίως δείχνοντας πολύ καλό χρονοδιάγραμμα να ε, νομοθετήσουν όταν αντιμετωπίζουν και όταν πρέπει να έρχονται σε επαφή επιχειρήσεις με τους καταναλωτές. Οι τεχνολογικές πτυχές προσθέτουν και άλλο χαρακτηριστικό περιπλοκότητας και γι' αυτό χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και είναι αρμοδιότητά μας να επεξεργαστούμε το κείμενο και δεν ξέρουμε όμω ποιε επιστημονικέ εξελίξει θα μπορούσαν μεσοπρόθεσμα να συμβούν. Δηλαδή εργαζόμαστε ε, επ' αυτού προσπαθώντας, ε, δουλεύουμε σήμερα, σκεφτούμε θα γίνει αύριο. μα, περιμένει πολλή δουλειά. Ε, θα ήθελα να εξετάσω τέσσερα βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα την προβληματική που καλούμε θα να βρούμε μια λύση. Οι διάφορε προβληματικέ είναι διαφορετικέ και η ισορροπία δεν είναι εύκολο να εξευρεθεί. Ε, λοιπόν, οι αρμοδιότητε η ΣΥΜΚΟ ΕΝΣΥΜΚΟ και θέλουμε να το και με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ΙΤΡΕ. Θέλουμε να έχουμε στενή συνεργασία μεταξύ των Επιτροπών επί τη ουσία επί συγκεκριμένων θεματικών τομέων. Στην ΙΜΚΟ θα πρέπει να συζητηθεί ει βάθο το μοντέλο διαδικτύου που θέλουμε. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε ε, το πώ θα γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων, μια συχνότητα, ε, με ποιε εξουσίε θα, θα πρέπει να δίνουμε αυτή την επεξεργασία ποια προβλήματα τίθενται, ποιε λύσει πρέπει να βρούμε. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και ο ρόλο των περίφημων cookies. Δηλαδή μπορούν ή μπορούν να μην ε, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο τη κυκλοφορία των στοιχείων. Ποια είναι τα όρια, ποιο είναι ο σκοπό τη χρήσεω. Ε, ποιες είναι, τι προσδοκίε έναντι των προσδοκιών που έχουν οι χρήστε για τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την προστασία τη ιδιωτική ζωή. Μετά είναι το θέμα συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτή τη Επιτροπή όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των data subjects και ε, πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά από τις επιχειρήσεις και στην εσωτερική αγορά και για τη μεταφορά των στοιχείων προς το εξωτερικό. Αναφερόμαστε και στις στοιχείες της προστασίας των καταναλωτών στην περίπτωση παραβιάσεως των, της χρήσης στοιχείων και την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να τροφοδοτεί ο καθένας ε, έναντι των ιστοσελίδων του διαδικτύου. Άρα συνδέεται αυτό πολύ στενά με αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως από τον συνάδελφο Πάμπλο. Ταυτόχρονο θα πρέπει να προσέξουμε και τα μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά. Ε, από πλευράς να δημιουργήσουν διακρίσεις όπως οι επενδύσει απευθείας από το εξωτερικό ε, και αυτό εντάσσεται και στο θέμα των πληρωμών. Και κάτι άλλο που συνδέεται με την εσωτερική αγορά ή με τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασία των δεδομένων και τι συνέπειε έχει αυτό για την προσέλκυση επενδύσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επαναπροώθηση τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Με αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη βεβαιότητα τη επιβολή του δικαίου και αυτό για προστασία των καταναλωτών. Αναφέρομαι στην επιλογή που αφορά τη λύση One Stop Shop αλλά και την κατανομή των ομοδιοτήτων και εξουσιών μεταξύ εθνικών αρχών ούτως ώστε η ερμηνεία του κανονισμού να μπορεί να είναι απόλυτα σαφής και να μην γίνει ένα εργαλείο marketing και πρόθεσης που δεν προστατεύει τον καταναλωτή. Ε, μια τελευταία πτυχή και την θέτω στην προσοχή σας είναι να πρέπει να σκεφτούμε και το online αλλά και τη ζωή, τη ζωή offline του κανονισμού που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πρώτα απ' όλα επικεντρώθηκα μέχρι τώρα επί του διαδικτύου αλλά ξέρω ότι παρά τις εξωτερικές ε, εμφανίσεις έχουμε και τον πραγματικό κόσμο πέρα από τον εικονικό που υπάρχει και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε και να το λαμβάνουμε υπόψη στην ανάλυση. Εκείνοι από εσά που ήδη έχουν εξοικειωθεί με την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν δει σε αυτά που είπα ότι θέλω να φτάσουμε σε βάθος, να αξιολογήσουμε την ουσία, να προχωρήσουμε ουσιαστικά, να πάρουμε αποφάσια το κείμενο. Ε, είμαι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ λεπτομερή εργασία βάθο, μαζί με του σκιώδει εισηγητέ. επίσης. Πολλοί από αυτούς είναι οι δυσκιώδει εισηγητέ, όπως για την τυποποίηση. Αυτό αν είναι καλός ιονός ευπρόσδεκτο. Ε, συνεργάστηκα με τον εισηγητή Άλμπερτ της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών και σίγουρα εμείς της Επιτροπή ΣΥΜΚΟ θα είμαστε πολύτιμη στήριξη αυτών, αλλά και η Επιτροπή Ελευθεριών θα είναι υποστηριχτής μας όσον αφορά ε, την διαμόρφωση και τον καθορισμό του τελικού κειμένου. Good. Um, can I just see who... Μάλιστα. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ, κύριος Αρίας, κυρία Γκάλο, η κυρία Κοράτσα Μπερίτ να αρχίσει και έχω και εγώ κάποια σχόλια μετά, γιατί είμαι ε, εν ενεργεία σκιώδης εισηγητής από την ομάδα μου. Θα είμαι σύντομη, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να ε, συνδυάσω και το τι γίνεται στη ΛΥΜΠΕ και, και το τι γίνεται στην δική μας επιτροπή. Υπάρχει το θέμα της αξιοπιστίας ε, των ε, επιχειρήσεων, ποιος είναι υπεύθυνο, να συλλέξει δεδομένα ε, και να τα αποθηκεύσει για πόσο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό, το ασφαλές ίντερνετ για τα παιδιά. Το συζητήσαμε και σε μια άλλη έκθεση, παιδιά και ψηφιακός χώρος ελπίζω να συμπεριληφθεί και αυτό και ε, στην ε, γνωμοδότηση της ε, εσωτερικής αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αν δει κανείς πόσα πράγματα προορίζονται για, τα παιδιά και είναι μάλιστα εν, εντελώς δυσανάλογοι με τα keywords που υπάρχουν για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα της υπεύθυνη ε, διαφήμισης και ένας αυτοπεριορισμός ε, στην ε, επιθετική διαφήμιση για τα παιδιά κάτω των 12 ετών, κάτι το, νομίζω ότι είναι πολύ, το οποίο είναι νομίζω πολύ σημαντικό και πρέπει να το βάλουμε στη γνωμοδότησή μας. Και το δικαίωμα της συγκατάθεσης είναι διαφορετικό πράγμα ο ενήλικας από το παιδί. το παιδί έχει πολύ λιγότερες δυνατότητες να δώσει τη συγκατάθεσή του το διαδίκτυο είναι πολύ σημαντικό ε, μέσο όμως και για τα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να τα προστατεύσουμε και για την ώρα θα σταματήσω εδώ. Μπορεί να είναι σύντομη τελικά η συζήτησή μας. Παύλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όχι, εγώ ήθελα λίγο να συνεχίσω αυτό που είπε η κυρία Κοράτσα. Εδώ είναι δύο θέματα. Το θέμα των παιδιών και των ανηλίκων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Το θέμα της εκπαίδευσης επίσης, διότι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε τώρα στο διαδίκτυο και που συνδέεται με το δικαίωμα στη λύθη. Τι σημαίνει αυτό. Κάποιοι έφηβοι γράφουν κάτι στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα. Ε, παράδειγμα, τι εννοώ ένας έφηβος βάζει μια προσωπική του πληροφορία που δεν τον πειράζει να το γράψει ως έφηβος, αλλά μπορεί να το πειράξει ε, πιο μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, όταν ελικιωθεί και είναι πολιτικός ή επαγγελματίας γενικότερα. Και το δικαίωμα στη λύθη υπάρχει και στο διαδίκτυο. Ε, και χωρίς νομοθεσία αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή μπορούν να σβήνονται και να χάνονται ή μένουν για πάντα. Και η διαπαιδαγώγηση για αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πρώτο που θα πρέπει να μαθαίνουν οι πιο νέοι είναι ε, όχι μόνο τα πλεονεκτήματα αλλά και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν στο διαδίκτυο. Αυτά προς το παρόν και θα κάνω μια τροπολογία για το δικαίωμα στη λύθη για την ανάρτηση προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα και αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει, γιατί δεν λειτουργεί αυτό το δικαίωμα στη λύθη, το να γράφω κάτι και να μετά να χάνεται, να το σβήνω, να μην μένει για πάντα. Ευχαριστώ. thank Ευχαριστώ πολύ. Μερικά σχόλια δικά μου τώρα. Αρκετά συνδέονται με αυτά που προανέφερα με τη συζήτηση του Παύλου Αρίας τη δουλειά που έκανα σαν εισηγητή για την ε, ηλεκτρονική προστασία, την προστασία σε ηλεκτρονικό επίπεδο της, της ιδιωτικής ζωής. Και αρκετέ πτυχές αναφέρθηκαν ήδη. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε ασχολείται με ένα θέμα, κυρίως οι πολίτες. Θέλουν αισθάνονται ότι τα στοιχεία τους προστατεύονται και είναι ασφαλή κυρίως τις οικονομικές συναλλαγές. Όμως θέλουν να μπορούν να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν αυτά σε κάποιες περιστάσεις επωφελής για αυτούς. Ίσως στα κοινωνικά δίκτυα, οικογενειακά δίκτυα, συναλλαγές. Θέλουν όμως να ελέγχουν τον τρόπο χρήσεώς τους. Βλέποντας αυτή την πρόταση, Νομίζω ότι αφορά προστασία. Δεν αναφέρεται όμως τον έλεγχο ή ελεγχόμενη χρήση των προσωπικών στοιχείων για συγκεκριμένους λόγους. Δεν τα αναφέρει αρκετά αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι πολίτες θέλουν να μπορούν να επιτρέψουν την χρήση των στοιχείων τους σε απόλυτα ελεγχόμενες καταστάσεις. Ο σκοπός για την οδηγία για τα cookies για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τα cookies. Δηλαδή, τα cookies αυτά, ηλεκτρονικοί μηχανισμοί επιτρέπουν να δουν ποια είναι η συμπεριφορά σου, παρακολουθούν τη συμπεριφορά σου στις σελίδες. Άρα η ιστοσελίδα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου, να τις αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται. Στην οδηγία την προστασία τη ιδιωτική ζωής στο διαδίκτυο ποια είναι μπορείς να συμφωνήσεις όταν είσαι ενήμερος. Όταν πας στην ιστοσελίδα, για πρώτη φορά σου βγαίνει ένα μήνυμα σχετικό. Στις καλές ιστοσελίδες ένα μήνυμα σου λέει ποια είναι η πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής σου ζωής και ποια η πολιτική τους για τα κούκις. Και ακόμα καλύτερες ιστοσελίδες δείχνουν ποια cookies χρησιμοποιούνται, πώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που μαζεύουν τα cookies. Άρα διαλέγεις τα καλά sites και αποφεύγεις αυτά που θεωρείς ότι μπορούν να παρακολουθούν τη δική σου ζωή. αυτό εννοούμε με έλεγχο. Και αφορούν αυτά και τη διαφάνεια. Δίνω τις πληροφορίες και μετά ελέγχω τι θέλω να κάνω. Και στο σελίδα, και το συνδέεται και με άλλα συναφή θέματα για την οδηγία του ηλεκτρονικού εμπορίου, πρέπει να μου δίνει στο σελίδα τη δυνατότητα να μπορώ να αλλάξω τι ρυθμίσει που έχω διαλέξει πριν οποιαδήποτε στιγμή θέλω. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή την οδηγία δεν βλέπω αυτή την πρακτική προσέγγιση εδώ. Ξεκινώντας από την αρχή μάλιστα. Κοιτάξτε τον ορισμό των προσωπικών στοιχείων. Λέει εσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με το υποκείμενο των στοιχείων. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που με αφορούν στη διάδρασή μου με στους σελίδες. Αλλά δεν ταυτίζονται με μένα. Και άλλες πληροφορίες που βρίσκονται εκεί ο αριθμός πινακίδων των αυτοκινήτων που έχω, σε βάση δεδομένων. Διότι αν θέλω να ψάξω να βρω μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και θέλω να ξέρω ποιο ήταν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτε, ίσω θέλω να ξέρω πού βρίσκεται στη χώρα και να ελέγξω κατά πόσο ισχύει το, η πινακίδα κυκλοφορία. Αυτέ οι εσδήποτε πληροφορίε με το υποκείμενο των πληροφοριών, τι σημαίνει αυτό είναι πολύ γενικόλογος νομικός ορισμός. Τόσο γενικόλογος που είναι ανέφικτο να εφαρμοστεί στην πράξη. Πώς θα αναλυθεί, πώς θα εφαρμοστεί. Και ίσως να είναι μια οδηγία που θα πρέπει να συνοδεύεται με, διάφορα, με διάφορες σημειώσεις και επεξηγήσεις και προσανατολισμούς για να καταλάβω τι εννοεί το κάθε σημείο. Ζητώ συγγνώμη που τον Τόμα Σέρτινγκ τη Γενική Διευθύνσεω για θέματα δικαιοσύνη δεν το συνέστησα πριν. Ε, Σα τον παρουσίασα. Η προσέγγιση με προβληματίζει. Αφορά κατά βάθο ε, την προστασία, αλλά δεν είναι τόσο καλά ε, ισορροπημένη και σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο για να παρέχει σωστά την προστασία. Χρειάζεται να μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη. Και δεν θα ικανοποιήσουμε απαραίτητε καταναλωτές καταναλωτέ αν δεν του επιτρέψουμε να καταλάβουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία τους και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία τους και πώς το ελέγχουν αυτό. Όσον αφορά την οδηγία για την προστασία τη ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο, είναι ένα καλό παράδειγμα εκεί πώς να βελτιώνεται μια φυστάμενη οδηγία. Οπότε, έρχομαι και σε ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται για μένα. Ε, μετά είναι το πιο ενδιαφέρον η κοινοποίηση παραβιάσεω ε, τη χρήση των στοιχείων. Όταν ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, με την κοινοποίηση για την παραβίαση των στοιχείων στην προστασία τη ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο, θέλαμε να βρεθούν λογικοί ορισμοί, πρακτικοί ε, ορισμοί στο πώ θα λειτουργήσει το σύστημα. Τώρα καταφθάνουν οι διάφορε, τα διάφορα Αυτό Το τη προτάσεω δεν σχετίζεται και πολύ με αυτά που κάναμε στην οδηγία την προστασία τη ιδιωτικής ζωή στον ηλεκτρονικό χώρο. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν ήταν η καλή εργασία που έκανε η Γενική Διεύθυνση για την ε, ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο. Η εμπειρία που είχαμε για την κοινοποίηση παραβιάσεως ε, των προσωπικών δεδομένων γιατί δεν εντάχθηκε εδώ ταχύτητα κοινοποίησεως, λόγοι κοινοποίησεως, σοβαρότητα της παραβιάσεως, όλοι οι άλλοι ορισμοί δεν εμφανίζονται εκτός αν κάνω λάθος. Άλλο, αναλογικότητα. Εγώ είμαι υπέρ κοινών κανόνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. και να μπορούν αυτοί που έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν σωστά τα στοιχεία. Το σύστημα πληροφοριών της εσωτερικής αγοράς που προαναφέραμε, που αφορά επικοινωνία μεταξύ των αρχών προστασίας των δεδομένων, είναι κάτι πρέπει να ισχύσει, να λειτουργήσει. Πρέπει να είμαστε σίγουροι θα γίνει. Το ξέρουμε καλά το θέμα. Όσο κινούμεθα προς cloud computing, όλο και περισσότερο, ποια πραγματικότητα διαμορφώνεται θα έχουμε marketing σε μια χώρα, επιχειρήσεις marketing, θα επεξεργάζονται τα στοιχεία μια εταιρεία που βρίσκονται σε άλλη χώρα τη ευρωπαϊκή Ένωση. και να συλλέγονται και στοιχεία σε τρίτη χώρα. Άρα θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποια δίκτυα. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο μηχανισμό. Γιατί? Να έχουν ένα σημείο επαφή εταιρείε. Για εκείνον που ελέγχει τα στοιχεία τη εταιρεία και που έρχεται σε επαφή με φορείς ελέγχου των στοιχείων σε διάφορες χώρες. Άρα ε, εργαλεία στοιχείων εσωτερικής αγοράς που θα αντιμετωπίζει και τα γλωσσικά προβλήματα που ίσως ανακύψουν. Και οι αρχέ προστασία των δεδομένων σε άλλες χώρες θα μπορούν να εξετάσουν περιπτώσεις παραβιάσεως ε, της χρήση των δεδομένων. προστασία των δεδομένων. Οι συγκεκριμένε απαιτήσει που επιβάλλονται σε εταιρείε, κυρίω στι μικρέ εταιρείε, και ενδεχόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές. Θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση οι εταιρείε να προσέχουν και να διαχειρίζονται σωστά τα δεδομένα. Όμως, αν είσαι μια μικρή εταιρεία και χρησιμοποιείς υπηρεσία cloud computing και όλο και περισσότερε εταιρείε το κάνουν αυτό και υπηρεσίε για επεξεργασία δεδομένων, cloud, σύστημα cloud κλπ. Και, και λογισμικού σε cloud, θα πρέπει να τις ενθαρρύνουμε να το κάνουν αυτό, διότι το ακούσατε πριν που συζητούσαμε την έξι του κ. Αρίας, που θέλουμε να προωθήσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτή η πρόταση λοιπόν πρέπει να διαφυλάσει τα στοιχεία χωρίς να εμποδίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς που αναπτύσσεται με νόμιμο τρόπο και να εξασφαλίζει ταυτόχρονα ότι εταιρείε που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να έχουν ιστοσελίδε όπου μπορούν να συλλέγουν στοιχεία από του ενδιαφερόμενου πελάτε που θέλουν να στείλουν τα στοιχεία και να έχουν επαφή μαζί του, να χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε cloud, μην ε, είναι είναι ανάλογο το κόστο και να φοβούνται για τι κυρώσει τόσο πολύ που να μην θέλουν να μπουν στην αγορά αυτή, την εσωτερική. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη έχει πετύχει τη σωστή ισορροπία. Και δεν ξέρω πόσο εξέτασαν αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή. Και ελπίζω ότι η κυρία Κόμη αυτό θα το θέσει στις συζητήσεις που συνεχίζονται διότι έχουμε μια καλή βάση, την έκθεση αυτή. Όμως, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μπει στο ψητό να δει το πώς ακριβώς θα αναπτυχθεί πρακτικά η ψηφιακή αγορά, πώς να ελέγχουν οι καταναλωτές πληροφορίες τους, πώς θα υπάρχει πρακτική ε, διάδραση με τις μελλοντικέ επιχείρησεις που θα λαμβάνουν χώρα χωρί να παρετούμεθα του γεγονότο ότι η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται με τρόπο που επεξεργάζεται κανεί ένα πολύτιμο αγαθό που δίνει ο καταναλωτή. Και τι θέλω να πω τώρα. Ότι αυτέ οι πληροφορίε είναι πολυτιμότατε για τι εταιρείε που θέλουν να τι χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, η επόμενη εξέλιξη όσον αφορά τα στοιχεία, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, και πάμε στο θέμα του ελέγχου τώρα, η επόμενη εξέλιξη θα είναι επιτρέπει στους πελάτες να εκμεταλλεύονται την αξία των στοιχείων τους που δίνουν στις εταιρείες με τρόπο που θέλουν οι πελάτες. Κάποιες δωρεάν υπηρεσίες που μας δίνουν πολλές ιστοσελίδες μηχανές ε, έρευνας ε, και εργαλεία χαρτογράφησης που είναι δωρεάν χρηματοδοτούνται από έσοδα διαφημιστικά κάποιο είδους και οι πελάτες έχουν τις υπηρεσίες αυτές δωρεάν. Κάποιοι πελάτες είναι ικανοποιημένοι με αυτή τη δωρεάν υπηρεσία. του αρέσει. Δεν ξέρω αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που είναι τόσο δυσδυτικό που αλλάζει όλο το εμπορικό μοντέλο στο οποίο βασιζόμαστε. Ίσως χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη συλλογή στοιχείων για διαφήμιση. Και έρχομαι στο θέμα του ελέγχου εκ νέου και τα στοιχεία των πελατών που είναι πολύ πολύτιμα και ίσω θέλουν να τα κρατήσουν εκτό αν έχουν καλύτερη υπηρεσία που του δίδεται και υπάρχει κάποιο κίνητρο να τα δώσουν. Δεν με νοιάζει αυτό. Έτσι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα. Αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι βλέπω ότι έχει, δοθ... ότι έχει αναλυθεί αυτό το θέμα. Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αλλάζει το εμπόριο, η αξία των στοιχείων. Δεν νομίζω ότι διατρέχει αυτή η ανάλυση την πρόταση. Καλή βάση μεν, Χρειάζεται πολύ βελτίωση δε. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Δεν ξέρω τώρα η κυρία Κόμη πώς θα αντιμετωπίσει το όλο ζήτημα. Θα δούμε. No. Okay. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως. Κύριε Ζέρντικ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που η Επιτροπή σας ε, βλέπει με τον ίδιο τρόπο τη σημασία και τη σπουδαιότητα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς. Έκανε τις προτάσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς και τα ακούσαμε για να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο ε, προστασίας νομικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον. Και πώς θα γίνει αυτό έχουμε ένα ενιαίο νομικό κείμενο που θα ισχύει ταυτόχρονα, κανονισμός δηλαδή, άμεσης εφαρμογής σε όλα τα κράτη-μέλη και έναν συνομιλητή ε, δηλαδή μία αρχή προστασίας δεδομένων. Αυτό λέγεται one-stop shop, μία ενιαία θηρίδα για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα θέλουμε να έχουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αλλά και μια πολλαπλώς ε, καλύτερη ε, προστασία για τα άτομα. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας πάντα ε, για διάλογο και πλήρη συνεργασία. Ε, μου επιτρέπετε να απαντήσω σε μερικά σημεία που ανέκυψαν ε, στην πορεία της συζήτησης. Οι δικές μας προτάσεις βασίζονται ιδίως σε ό,τι αφορά τους ορισμούς, στα όσα ορίζει το άρθρο 8 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ατομικά και προσωπικά δεδομένα, το άρθρο 16 της συνθήκης και ιδιαίτερα υπάρχει μια οδηγία 95 ε, κάθετο 46 που ισχύει γενικά για την προστασία των δεδομένων και έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχή στην πράξη. Ε, και offline και online, λέει η συγγήτρια. Δεν πρόκειται μόνο για το διαδίκτυο, δεν πρόκειται για τα cookies, πρόκειται και για την πραγματική ζωή, την καθημερινή ουσιαστική ζωή σε κάθε της ψυχή και γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, μια γενική μορφή κανονισμού. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι Έχουμε πολλά μέσα ε, στα νομοθετικά κείμενα για να αυξήσουμε τη διαφάνεια και υπάρχει μια ρητή αρχή διαφάνειας την οποία εισάγουμε τώρα που δεν υπήρχε στο παρελθόν υποχρέωση ενημέρωσης, πληροφόρησης ακριβώς για να έχει ο κάθε ε, άνθρωπος πολύ μεγαλύτερο έλεγχο για τα ίδια του τα προσωπικά δεδομένα. Η ε, υποχρέωση τροποποίησης των στοιχείων, των προσωπικών δεδομένων, το ξέρουμε και σήμερα στην οδηγία για την ιδιωτική ζωή. Με εκπλήσει πάρα πολύ αυτό που λέτε, διότι κατά την άποψή μας έχουμε πετύχει 100% συνέπεια. Αλλαγές στο κείμενο γίνονται κυρίως και μόνο λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για πρόταση κανονισμού. Και βεβαίως χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερες διατάξεις και οδηγίες ε, εφαρμογή σε σχέση με ένα νομικό κείμενο που να είναι οδηγία. Ε, εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλαμε πολλές προσπάθειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δούμε πού ενδεχομένως ε, μπορούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και πού ενδεχομένως μπορούμε να μειώσουμε τις υποχρεώσεις που θα επιβαρύνουν τις μικρομεσαίες στην καθημερινή μας πρακτική εμείς συναντούμε ένα άλλο επιχείρημα, ότι έχουμε δημιουργήσει υπερβολικές ε, σε αριθμό εξαιρέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε για την προστασία ε, ενός θεμελιώδου δικαιώματος δεν μπορούμε να έχουμε καμία δικαιολογία για τόσες εξαιρέσεις. Οπότε μάλλον βρισκόμαστε στη μέση με τις προτάσεις που κάνουμε. Αυτά από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρόμαστε για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για ενημέρωση και ό,τι άλλο θέλετε διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Could Μήπως μπορείτε να πείτε για την οδηγία ε, περί προστασίας του ιδιωτικού βίου ορισμένα πράγματα και τη σχέση της με αυτό που συζητάμε. Προβλέπουν οι προτάσεις ακριβώς λόγω του, αλλά, ε, της αλλαγής του 2009 ε, δεν ασχολούμαστε με αυτό. Αυτό που λέει η μερίσια διάταξη μάλλον το πω ε, μπορεί να υπάρχουν επικαλύψεις και για να μην υπάρχουν επικαλύψεις θέλουμε ε, στην κοινοποίηση ε, των στοιχείων να υπάρχει υποχρέωση ε, αναφοράς. Σε καμία περίπτωση δεν διαφέρουν οι νέες προτάσεις σε σχέση με την πρόταση για το privacy, την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Θέλουμε ακριβώς να αποφύγουμε αυτό, να υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις και κανόνες. Τα βλέπουμε ίσως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά θα το εξετάσουμε. Κύριε, Κόμη ή οποιοδήποτε άλλο θέλει να πάρει το λόγο πριν. Αυτό είναι και ένα από τα σημεία που θα λάβουμε υπόψη και θα επιφέρουμε περισσότερες διευκρινήσεις επί η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Εγώ θα ενημερώσω και για τις πρόσφατες σκέψεις και για τα πρόσφατα ερωτηματικά που θα βγουν και τις άλλες επιτροπές. Θα σας ενημερώσω, θα συνεργαστούμε λοιπόν σε επόμενες συνεδριάσεις και σε επόμενες συναντήσεις Βέβαια έχουμε τη μέγιστη ε, διαθεσιμότητα για να ακούσουμε τη συνεισφορά όλων και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. να πείτε ορισμένα πράγματα για το χρονοδιάγραμμα ίσως. Ε, ε, Κοιτάξτε. Περιμένουμε για το χρονοδιάγραμμα μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών θα έλεγα ότι ενώ βλέποντας το χρονοδιάγραμμα τη Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που μιλάει ψηφορία του χρόνου το Μάρτιο, αν ισχύει αυτό, περί αυτού πρόκειται. Απάντηση. Ναι, στην ΙΜΚΟ τον Ιανουάριο και λίγο πολύ οι προβλέψεις που είχαμε δει μπορείτε να τις επιβεβαιώσετε, ξεκριβώσετε μετά τη συνεδρίαση 21 Ιουνίου ανταλλαγή απόψεων που έγινε σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2012 το σχέδιο εκθέσεως, παρουσίαση αυτού, συζήτηση ο δύο εκθέσεως της 11 Οκτωβρίου, προθεσμία υποβολή τροπολογιών 6 Νοεμβρίου, ανταλλαγή απόψεων οι τροπολογίες συζήτηση 29 Νοεμβρίου, συζήτηση των συμβιβαστικών 17 Δεκεμβρίου, ψηφορία στην ΙΜΚΟ 24 Ιανουαρίου. Και υπάρχει και αυτό μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα και τι αποφάσει θα πάρετε κι εσεί, γιατί είναι work in progress. Συνεχίζονται εργασίε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να φέρω πιο κοντά, τη, να συντομεύσω το χρονοδιάγραμμα τη Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Έχετε δίκιο, μα δίνει περισσότερο χρόνο. Αντίθετα, αυτοί θα θέλουν να αναβάλουν. Θέλουν να αναβάλουν, ε. Καλώ λέει ο Πρόεδρο. Θέλουν να κάνουν πολλέ αλλαγέ και βελτιώσει από ό,τι ακούεται αυτή η περίπτωση, έτσι. Καλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μας ε, ενημερώνετε σχετικά με εργασίας Επιτροπής ε, Ελευθεριών ανεξάρτητα της συζήτηση για διευρυμένη συνεργασία ή κάποια στοιχεία που θα αφορά τα στοιχεία της ενιαίας αγοράς όλα αυτά πρέπει να παρακολουθούμε τις εργασίες τους κυρίως αν ετοιμάζουν ακροάσεις, σεμινάρια, ό,τι ετοιμάζουν. Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν έχουμε τόσο χρόνο όσο νόμιζα ναι. τελικά. Έχει περάσει, ο χρόνο, έχει περάσει η ώρα, πω Συγγνώμη, εγώ φταίω. Uh, Με είχε τόσο απορροφήσει αυτό το θέμα τη προστασία δεδομένων. Τέλο πάντων, είναι εδώ η κυρία Γκάλο και θα μα μιλήσει για, τα για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών. Ε, είναι συντάκτη νομοδότηση ε, για την έκθεση τη Επιτροπή Βιομηχανία. Ε, ο κύριο Σμιτ δεν είναι εδώ, η κυρία Ρούλε δεν είναι εδώ. Εγώ όμω είμαι εδώ, οπότε δύο σκιώδεις είναι εδώ. Ο κύριος Φιλίππο Μινιστέρ είναι εδώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σωστά. Ναι, υπάρχει εδώ κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι εγώ. Ποιο είναι το όνομά σας όμως. Μάρτιν Νιούμπελερ. Ε, από την ε, DG Connect. Θα γίνει σύντομα DG Connect η ε, γενική μας διεύθυνση. Όχι ακόμα όμως. Μάλιστα, ναι. Σύντομα DG Connect, λοιπόν. Προσεχώς. Κυρία Γκάλο, θέλετε να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καταλαβαίνω το γεγονός ότι σας προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό το θέμα της προστασίας δεδομένων ε, και λιγότερο με αυτό το θέμα σας απασχολεί, το θέμα των ε, διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών. Κυρίως όταν το, το σχέδιο κανονισμού που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα καλό κείμενο και συνεπώς ε, δεν ε, χρειάζεται ιδιαίτερες ε, τροποποιήσεις, μόνο ελάχιστης σημασίας. Η πρόταση δίνει προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και προτείνει στόχους και προτεραιότητες για κοινά σχέδια με σκοπό να μην υπάρχουν ε, ε, σημεία συμφόρησης. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό ε, με την διασύνδεση στα δίκτυα και την διασυνοριακή πρόσβαση σε δημόσιες ψηφιακές υποδομές. Στο σχέδιο γνωμοδότησής μου επιμένω ιδιαιτέρως σε τρία σημεία Πρώτον, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δράσει εκεί όπου υπάρχουν αδυναμίες στην αγορά και ε, όπου έχουν εντοπιστεί. Για να ενισχύσει τη συνοχή της επικράτειάς της, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει ακόμη και οι πιο αραιοκατοικημένες περιοχές, οι πιο απομονωμένες περιοχές έχουν μία πρόσβαση καλής ποιότητας στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Έχω λοιπόν υποβάλει δύο τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, θα ήθελα, ήθελα να επιμείνω στην αναγκαιότητα υποδομών ε, τηλεπικοινωνιών αποτελεσματικών ε, με τη διεύρυνση του φάσματων ε, νέων ε, συσκευών όπως τα tablets, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα κλπ. Και τρίτον, μου φάνηκε σημαντικό να τονίσω ότι ένας από τους στόχους ε, των ε, ε, σχεδίων κοινή ωφέλεια είναι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, που επιζητούν υψηλή ταχύτητα, γιατί είναι ανεπαρκής η ταχύτητα και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος ε, γιατί η υψηλή ζήτηση είναι αυτή που θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ε, που θα απευθύνονται στους καταναλωτές. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε το είχε διαπιστώσει νωρίτερα στην αιτιολογική της έκθεση αλλά δεν το μετέγραψε με πάρα πολύ σαφή τρόπο στο διατακτικό του κανονισμού. Επομένως, Αυτά ήταν τα σημαντικότερα που ήθελα να πω και ελπίζω ότι το κείμενο αυτό με αυτό το νέο μηχανισμό διασύνδεσης θα ε, ενθαρρύνει μια νέα δυναμική για ε, την υλοποίηση αυτής της ε, ψηφιακής ε, αγοράς και περιμένω βεβαίως με μεγάλη αγωνία τα σχόλια των συναδέλφων μου που είναι πάρα πολύ απασχολημένοι και δεν με ακούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σφίτς. Σίβιετς. δεν ξέρω αν το είπα καλά το όνομά σας. Σίβιετς. Σίβιετς. Πλησιάζεται, πλησιάζεται στην τέλεια προφορά. Κάνω ό,τι μπορώ, λέει ο πρόεδρος. Έχω έναν ολόκληρο κατάλογο ε, των ε, ε, ανθρώπων που έχουν προφέρει λάθος το όνομά μου και δεν είστε στον τελευταίο, στην τελευταία θέση του καταλόγου αυτού. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, την χάνει να δημιουργείται η εντύπωση ότι το θέμα δεν είναι σημαντικό επειδή είμαστε τόσο λίγοι παρόντες. Παρ' όλα αυτά, εάν κοιτάξουμε τι συμβαίνει σήμερα, ακριβώς σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνδέεται με αυτές τις δύο απλές λέξεις, διαδίκτυο και ψηφιακό, θα καταλάβουμε ότι αυτό που συζητούμε έχει ύψιστη σημασία. Για το λόγο αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να τονίσω ότι εδώ η Επιτροπή μας ονομάζεται Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Ε, και για το θέμα αυτό θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ξεκάθαρη άποψη και κατηγορηματική. Σε τέτοιους καιρούς είναι ζωτική σημασίας να ε, εγκρίνουμε αυτή την νομοθεσία. Σήμερα η πρόσβαση, για να μην πω η μη πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι κάτι ε, από το οποίο εξαρτάται η ένταξη ή ο αποκλεισμό. Όπως ήταν παλαιότερα στην κοινωνία μας, σε παλαιότερους αιώνες, η εκπαίδευση, η παιδεία. Μερικοί θα σας πούν ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι μέχρι και ανθρώπινο δικαίωμα γιατί είναι απαραίτητη για να φέρει την πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη. Ορισμένοι θα σας πούν ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου είναι ε, η προϋπόθεση ίδια για να ξεπεράσουμε την κρίση. Τέτοια σημασία έχουν αυτά. Οπότε, αν μιλήσουμε για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα δικαιώματα αυτά δεν θα γίνουν ποτέ σεβαστά εάν δεν έχουμε ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών που να λειτουργεί με σωστό τρόπο και να έχουμε ελεύθερη διαβίβαση δεδομένων, Και πώς θα γίνει δηλαδή τώρα να ε, απελευθερωθεί όλο αυτό το δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα έγγραφο για τις τρίτες χώρες που ορίζει ότι η έλλειψη της πρόσβασης στο διαδίκτυο ε, αποτελεί κίνδυνο για την ελευθερία την ίδια. Δηλαδή, αν εμείς δεν καταφέρουμε να εγγυηθούμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν διασυνοριακή ε, μεταβίβαση ή διαβίβαση των δεδομένων μέσα σε ένα δίκτυο, Εάν δεν καταφέρουμε να βοηθήσουμε προς την ανάπτυξη αυτό θα υπονομεύσει όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την ίδια την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών και άλλα τεινά. Γι' αυτό το λόγο προσωπικά Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Κάποιος μη ειδικό θα πει ότι καλά συζητάτε για καλώδια, για σύρματα, για ασύρματα για πρόσβαση στο διαδικτύο. Όχι, δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για τον πολιτισμό και για οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι τεχνικό το ζήτημα. Η ε, ανάπτυξη ε, των δικτύων που αναφέρεται σε αυτό το κείμενο είναι η ίδια προϋπόθεση για την επιτυχία. Ακόμα και αν δεν είναι πολύ δημοφιλής αυτή η έκθεση. Χωρίς ταχεία διαβίβαση των δεδομένων ε, θα χάσουμε το τρένο της πρόοδου, θα μείνουμε πίσω και ε, μπορώ να σας πω ότι τελικά θα καταντήσουμε να οπισθοδρομούμε. Θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τη σημασία του θέματος. Δεν είναι τεχνικό το θέμα, είναι θέμα πολιτισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιβίτς. Thank you. Um, just some comments from me as the... Και κάποια σχόλια εγώ θα ήθελα να κάνω. Συμφωνώ. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό, ε, ένας πολύ σημαντικός τρόπος για να επιτύχουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο περιοριστικό το κείμενο όσον αφορά τα σχέδια κοινή ωφέλεια δεδομένων των ε, αλλαγών που λαμβάνουν χώρα υπονοεί ό,τι αφορά τα τηλεπικοινωνιακά διευρωπαϊκά δίκτυα, όμως ε, αφορά πολύ περισσότερα πράγματα. Μιλάμε, ας πούμε, για το, ε, τη γραμμή βοήθειας για την ασφάλεια των παιδιών. Λέει επίσης ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με τις, ε, την ύπαρξη των συγκεκριμένων προδιαγραφών όμως δεν ξέρω αν είναι απλώς ένας περιορισμός αυτά που αναφέρονται εδώ επιγραμματικά, όπως για παράδειγμα η ευφυή ενέργεια ή αν ε, είναι απλώς ένα παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται. Και υπ' αυτήν την έννοια... Ε, ελπίζω να μην αλληλεπικαλύπτεται ή να μην περιορίζει κάποιες άλλες πτυχές. Υπάρχουν κάποια γενικά κριτήρια που αναφέρονται εδώ και το παράρτημα είναι κατά τη γνώμη μου πολύ διεξοδικό, πολύ περιοριστικό και η κυρία Γκάλο πρέπει να το εξετάσει αυτό, να το διερευνήσει. Αναφέρεται εδώ Τονίζεται μάλιστα ότι η χρηματοδότηση μπορεί να υποστηρίξει σχέδια τα οποία έχουμε ήδη αναγνωρίσει όπως διαρθρωτικά κονδύλια για ζητήματα ανταγωνιστικότητας ε, ε, ή μιλούμε και για εμπορικές ε, συναλλαγές. Παρατήρησα για παράδειγμα ότι κάποιον κάποιος από τον προγραμματισμό ε, για την ανάπτυξη μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, όμως η πληρωματική χρηματοδότηση αφορά ε, την, ε, την υποδομή του υλικού καταρχάς και αυτό είναι τεράστια ε, χρηματοδότηση ε, που ε, θα αφορά πολύ ευρύτερα προγράμματα, πολύ μεγαλύτερα. Και μου φαίνεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, οι ευρυζωνικές οι ασύρματες ευρυζωνικές, τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα ε, είναι ε, μεν πολύ σημαντικά για όλες τις περιοχές, όμως πρέπει να υπάρχει και μία ε, τεχνολογική ουδετερότητα. Αυτό είναι κάτι που εμένα με ικανοποιεί. Θα υποβάλω κάποιες σχετικές τροπολογίες. Κυρία Ρούλε, ήρθατε, θέλετε να πάρετε το λόγο, γιατί είστε και σκιώδης Α, όχι. Δεν είστε εσείς συνάδελφος Έγκστρομ. Αυτά είχα να πω εγώ. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κάτι να μας πει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, την ε, κυρία Γκάλο για την έκθεσή της ε, και τους σκιώδεις εισηγητές. Η έκθεση αναφέρεται στη σημασία του cloud computing νέων υπηρεσιών, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι μια αξιολόγηση που βρίσκει σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η έκθεση αναφέρει επίσης τη σημασία της διασύνδεσης των ε, περιοχών της υπαίθρου, των πιο αεροκατοικημένων περιοχών ή των ε, οικονομικά λιγότερο ευημερουσών περιοχών και το συνδέει επίσης και με την ψηφιακή ενιαία αγορά που είναι επίσης μία από τις προτεραιότητες του προγράμματος που προτείνουμε. Ένα σχόλιο αφορούσε την προσφορά και τη ζήτηση και η κυρία Γκάλο ήθελε να δημιουργήσει έναν ενάρετο και όχι φαύλο κύκλο. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε και ελπίζουμε ότι το καταστήσαμε παρκώς σαφώς στην πρότασή μας ότι καλύπτει δύο βασικές πτυχές. Η πρώτη είναι τα προγράμματα τα ευρυζωνικά που είναι ε, η προσφορά και από την άλλη είναι η διαλειτουργικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ε, online ε, ή υποδομές οι ψηφιακές που ελπίζουμε ότι θα ενθαρρύνουν στην ψηφιακή ενιαία αγορά τη ζήτηση. Ελπίζουμε λοιπόν να συνεισφέρουμε και εμείς αυτόν τον ενάρετο κύκλο της προσφοράς και της ζήτησης. Όσον αφορά τώρα τον περιοριστικό χαρακτήρα του παραρτήματος. Ναι, είναι τεχνολογικό ουδέτερα τα προγράμματα όσον αφορά την, τα, την ευρεία ζώνη. Όντως τα ασύρματα ε, συμπεριλαμβάνονται το βασικό κριτήριο για τις τεχνολογίες που, πρέπει να, που μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι η ταχύτητα ε, μετάδοσης, ε, που είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ, σημαντικό πλαίσιο στο, είναι πολύ στο πλαίσιο της ψηφιακής ατζέντα. Θέλουμε 30 ε, bit ε, για κάθε πολίτη. Οπότε θα δούμε το αποτέλεσμα και για τους ε, καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Τώρα, η σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα. Ε, Πρόεδρε, αναφέρατε το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Το δεύτερο τμήμα της πρότασης, ε, το θέμα των ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών και το διασυνοριακότητα αυτών, έχει άμεση σχέση με το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και κοινοτομία. Κάποιες από τις ε, σχετικές ε, ε, δράσεις αναπτύχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν ε, από το κοινό, ε, από το ε, CIP, από το πρόγραμμα αυτό για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και πρέπει να βρούμε τώρα τεχνικές λύσεις σε ορισμένα προβλήματα, να υπάρξουν λύσεις οι οποίες μπορούν να είναι αποδεκτές από νομικής και διοικητικής απόψεως από τις αρχές τις εμπλεκόμενες, γιατί μιλούμε κυρίως εδώ για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αλλά όχι μόνο για αυτό το θέμα. Τώρα, διαρθρωτικά ταμεία. Κυρίως ε, στα προγράμματα τα ευρυζωνικά ε, θεωρούμε ότι μπορούν να επισέλθουν τα ε, κονδύλια αυτά για τα project bonds, για τις για, τις, ε, για τα δάνεια μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για τα προγράμματα τα οποία δεν είναι αρκετά βιώσιμα ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τέτοιο τρόπο. Μία λύση για αυτά θα ήταν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία συμπληρωματικά για να υπάρχει αρκετό κεφάλαιο ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν ε, από την ε, τράπεζα τα ε, προγράμματα αυτά. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τις αφήσεις σας Κυρία Γκάλο, θέλετε να συνοψίσετε. Να συνοψίσω όχι ακόμα, γιατί δεν ολοκληρώνουμε, το χρονοδιάγραμμα ίσως αν όχι στους συναδέλφους, τους ε, βοηθούς τους που παρευρίσκονται. Προθεσμία για τις τροπολογίες 29 Ιουνίου, εξέταση των τροπολογιών 18 Σεπτεμβρίου και ψήφιση της έκθεσης ε, καταρχήν ε, στις 11 Οκτωβρίου. Είναι λογικές προθεσμίες και μπορούμε να τις στηρίσουμε. Ιδιαίτερα αν έρθουν γρήγορα οι τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Good. Well, thank you. Καλώ. ευχαριστώ πολύ όλου σα. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του σκιώδει εισηγητέ και εισηγήτριε. Ολοκληρώνεται εδώ η απόψηνη υπογευματινή συνεδρίαση. Στις 5 συνεδριάζουν οι συντονιστέ. Γιατί έχουμε να συμφωνήσουμε μερικά άμεσα ζητήματα προς διεκπαιρέωση. Ευχαριστώ πολύ και χαίρετε. Ε, αποχαιρετώ και τους ακροατές μας στο διαδίκτυο και θυμίζω ότι έχουμε νέα έκδοση ε, του newsletter. Αν θέλετε να εγγραφείτε πρέπει να πάτε στην ιστοσελίδα μας και θα σας στέλνουμε τακτικά ένα αντίγραφο των νέων του δελτίου της Επιτροπής μας. Και μπορείτε μέχρι να γίνετε και φίλοι της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο.